και φυσικά εναπόκειται στην, ε, στο Ευρωπαϊκό, στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να διακριβώσει αν οι κανόνε τη ομάδα η συνάδουν με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα το αποφασίσει η συνέλευση των πρόεδρων. Έχουμε το ε, χρονοδιάγραμμα των περιόδων ολομέλειας για το 2014 που έχουν ε, γίνει δεκτές από τη συνέλευση των Προέδρων η Τετάρτη 12 Ιουνίου στι 11.30 Συγγνώμη, η Τρίτη 11 Ιουνίου στις 12 είναι η προθεσμία για τροπολογίε και η ψηφοφορία θα γίνει την επόμενη μέρα Τετάρτη στι 11.30. Βάσει του άρθρου 47 μας με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού 74 συγγνώμη, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έχουμε, την Τετάρτη θα υπογράψω 10 κείμενα τα οποία έχουν γίνει δεκτά βάσει της ε, νομοθετη... κανονικής νομοθετικής διαδικασίας. Θα δημοσιευτούν στα πρακτικά αυτή τη Ολομέλειας τα κείμενα των νομοθετημάτων αυτών. Ερχόμαι τώρα στο σχέδιο εργασιών για αυτή τη βδομάδα. Καταρχήν για σήμερα υπάρχουν προτάσεις αλλαγής ημέρησης διαταξία σήμερα.